σε κάποιες ανακοινώσεις. Η κυρία Ούλα Τούρνες ε, έγινε μέλος της ε, κυβέρνησης της Δανίας. Να τη συγχαρούμε για τον ε, διορισμό της. Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι η έδρα της χειρεύει από 29 Φεβρουαρίου 2016. Από τις